Okay, everyone, hello. Let's start the voting session. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και καλώς ορίσατε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Αν δεν θέλετε, παρακαλώ να ψηφίσετε όρθιοι, καθίστε. Αλλά τουλάχιστον προετοιμάστε τον... την κάρτα ψηφοφορία σας για τις πρώτες εκθέσεις θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τις κάρτες σας παρακαλώ. Πολύ ωραία πρώτη ψηφοφορία. Για τις ε, εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα από βαρέα οχήματα και ψηφίζουμε στη συμφωνία πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη. And it is closed. Εγκρίνεται. Δεύτερο θέμα. Ένσταση. Για την εμπορία τροφίμων και ζωοτροφών από γενετικά τροποποιημένα ζαχαρότευλα 7 7-1. Ψηφίζουμε επί της ένστασης. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκ νέου, μια ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 για τα ανώτατα όρια για μια σειρά ουσιών εντός και επί ορισμένων προϊόντων. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. question. Okay, now we vote on Μάλιστα, και τώρα ψηφίζουμε ε, επί μια προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του πακέτου κυκλική οικονομία σε ό,τι αφορά τα χημικά προϊόντα και τη σχετική νομοθεσία για τα απορρίμματα. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για το ίδιο θέμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε επί μιας άλλης προφορικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία της Ευρω... Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς κατά των ε, αρνητικών συνεπειών σε ό,τι αφορά τα ζώα στην Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Για το ίδιο θέμα, προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. να ψηφίσουμε πια μια έκθεση πρωτοβουλία για την εφαρμογή τη οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, eco-design. Ψηφίζουμε την τροπολογία, τη συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχέ, ε, ε, εγκρίνεται. Η 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία βαριθμών 91. Ψηφίζουμε. Είσαστε κατά, κύριε Χερμπλάντε. Πέρασα. Με τον κύριο Χερμπλάντη εξακολουθεί να εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 104. Ψηφίζουμε. Για την 104. Κύριε Χερμπράντη, καταψηφίζετε. Πέρας. Δεν τα καταφέραμε αυτή τη φορά. Στον κύριο Χερμπράντη το λέω. Εγκρίνεται η τροπολογία. Μπράβο Μαρκρέτ. Ήτρε έξι. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίβεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Έλεγχος την 127 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρασε Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ε, εντάξει. 129 ψηφίζουμε παρακαλώ να δούμε ποιοι ψηφίζουν υπέρ, ποιοι κατά. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Μήπω όντω απορρίπτεται. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Λουδικά. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 και 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137. Έλεγχος για την 136 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Οι πράσινοι με δυσκολεύουν κάπως σήμερα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. 137 και 140. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Δεν τολμώ να αποφασίσω πλέον από μόνη μου. Πέρας. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 310 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την ήτρε 10. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήτρε 11. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την ΙΤΡΕ 11. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 194. Πέρας. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει. Μάλιστα καταπίπτει. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος παρακαλώ για την 4. Ψηφίζουμε. Το καταλάβω. Απορρίπτεται. Ο κύριος Χερμπράντη τώρα πια έχει την κάρτα του μαζί. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επτά 12 και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε, ας ξαναδούμε την... Όχι δεν πειράζει, ας κοιτάξουμε ηλεκτρονικά την νέα έναρξη. Και πέρασε. Εγκρίθηκε. Η 11 και 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ τον 28. Πέρας. Έγκρινεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 36 πέρας εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 και 40 υπέρ Κατά. Έλεγχος παρακαλώ τις 39 και 40. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε α, υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήτρε β και σ. Ήτρε μάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήτρε E υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήτρε f υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Και αυτό ήταν. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Now. Και τώρα ψηφίζουμε για την πολιτική συνοχή και την κυκλική οικονομία. Έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. Συμβαστική 1. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά έλεγχος για την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε για την 27 ωστόσο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ,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 Δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Σαν να συμφωνήσετε πάλι όλοι. 47 υπέρ, ωραία, εγκρίθηκε. 48 υπέρ, κατά. Από, να ελέγξουμε για το 48. Εγκρίνεται 49 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Πέρας, εγκρίθηκε. έκθεση ιδέας πρωτοβουλία κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνας. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές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 εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρώτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τετάρτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται αυτή.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 Τώρα περνάμε στο σε σημείο 19, το μέλλον των τροφίμων της Γεωργίας. Συμβαστική 1, ε, συμβαστική συγγνώμη, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Χάθηκε στα χρώματα, λέει η πρόεδρος. Που πάμε, 13, συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολλές σελίδες πιο κάτω, 137 λέει πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 142 πέρας απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 145 Έχει αλλάξει η αριθμίση από ό,τι φαίνεται. Πέρας της ψηφορίας. Υπέρ. 146 υπέρ κατά 146. 145 146. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 153 επέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τα 153 άρχεται πέρας απορρίπτεται το είχατε παρατηρήσει λέει πρόεδρος συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές Θα ψηφίσουμε για 165 ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν ήμασταν τελικά υπερικατά. Ψηφίσουμε για 165. Για 165. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τα 173 πέρας εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, λέει πρόεδρος, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα αποτέλεσμα. Πέρας της ηλεκτρονικής, γιατί 181 εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. κατά 17 ήταν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 199 υπέρ κατά 199 και πάλι υπέρ εγκρίνεται λέει πρόεδρος 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές που είναι η λέει πρόεδρος 239 υπέρ οπότε εγκρίνεται 240 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 240 πέρας Εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, ο πρόεδρος. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Uh, you have noticed here. Yeah. Θα δείτε ότι έχουμε μια καταπίπτη τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, 5 και 6 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 7 κατά πίπτη, 8 και 9 μαζί. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 και 13 μαζί. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Για τις 12 και 13. 12 και 13 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. And it is closed. Πέρας. Εγκρίνονται. Δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Τουλάχιστον δύο ομάδες δεν είπαν τίποτα. Δεκατρία υπέρ κατά άποχες έχουμε και εποχές 13 13 άρχεται ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Πέρας εγκρίνεται η 13 15 λέει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 18 The vote is Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 18 19 υπέρ Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 19. It's Περάς. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για την 20. Ποιος είναι υπέρ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 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 41 It's closed. Περάς εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 66. It's closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81. Όχι, καλά, προς συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 102 άρχεται πέρας εγκρίνεται 113 υπέρ κατά 113 υπέρ ξαναλέει η πρόεδρος κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψήφος ή ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το σύνολο άρχεται It's closed Πέρας. Εγκρίνεται. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ψηφίσουμε για τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 5 λέει πρόεδρος. 5, έτσι. Όλοι ψήφισατε υπέρ, έτσι δεν είναι. Έξι. Όχι έξι λέει πρώτος, εφτά. Εφτά. Εφτά ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οχτώ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δέκα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος ηλεκτρονικά. Άρχεται. And και εγκρίνεται. Ποιος καταψήφισε? Αυτά. τελειώσαμε τις πληροφορίες και με τη συνεδρίασή μας. Οπότε εύχομαι σε όλους σας ένα καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9 και έχουμε και τον Επίτροπο με την ομοθεσία για τα τρόφιμα. Πολύ ενδιαφέρον.